Συνεχίζουμε την ημερήσια διάταξη με την εισήγηση Λάμστορφ ε, για ε, το θέμα των προσφυγών για τα θέματα άμενας και ασφάλειας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Υπάρχουν 13 αποστολές της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκή Ένωση, ανά τον κόσμο. Εννέα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Σε τέσσερις από αυτές συμμετέχουν και στρατιωτικέ δυνάμει των χωρών μα, ορισμένε φορέ αστυνομικέ δυνάμει, σε δύσκολε συνθήκε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πολλέ άλλε αιστείε κρίσεων και ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση ε, ευρωπαϊκών παρεμβάσεων, η οποία δεν πρόκειται να μειωθεί. Γνωρίζουμε επίση ότι εμεί οι Ευρωπαίοι συχνά δεν είμαστε σε θέση να εκτελέσουμε τι αποστολέ μα όπω θα έπρεπε. Με με άριστο εξοπλισμό, διαλειτουργικό και με ε, ε, στρατηγικό βάθος. Οφείλουμε να τα επιτύχουμε αυτά, διότι τα χρωστάμε και στους σταθιωτικούς μας και στους αστυνομικούς μας, οι οποίοι ε, ε, δραστηριοποιούνται σε αυτές ε, τις αποστολές. Και πρέπει να το κάνουμε. Αλλά δυστυχώς είναι κατακαιρματισμένη η αγορά μας. Οι 27 μας χώρες μέλη έχουν 90 σχεδόν διαφορετικά προγράμματα έρευνας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μόνο 27. Έχουμε και σημαντική απόσταση των ε, προμηθευτών, με τους λεγόμενους ιστορικούς προμηθευτές που δεν είναι πάντοτε οι καλύτεροι στον, ε, στην ευρωπαϊκή αγορά εξοπλισμών κινούνται 91 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο 13% ε, γίνονται προσκλήσεις εκτός ενδιαφέροντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και η Γερμανία είναι μάλιστα ουραγός με 2 μόνο οι ένοπλες δυνάμεις μας λοιπόν δεν διαθέτουν τον καλύτερο εξοπλισμό και τα χρήματα των φορολογουμένων κατασπαταλώνται. Ο εξοπλισμός γίνεται όλο και ακριβότερος, όλο και δαπανηρότερος. Οι δε αμυντικοί εξοπλισμοί μειώνονται. Είναι προφανές λοιπόν περί τίνο πρόκειται. Δεν ζητούμε περισσότερες αμυντικές δαπάνες. Ζητούμε τα χρήματα που ήδη υπάρχουν και διατίθενται να δαπανώνται με καλύτερο και ευφιέστερο τρόπο. Αυτό το οφείλουμε και στους φορολογουμένους μας. Ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε έκθεσή του έχει ζητήσει να καταθέσει οδηγία, σχέδιο οδηγία για ε, το θέμα αυτό. Και το έπραξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για μένα ως εισηγητή ήταν σημαντικό ότι ο πρόεδρος Σαρκοζή, ε, ε, μιλώντας για τις προγραμματικές δηλώσεις της Γαλλικής Προεδρίας, τόνισε και το θέμα αυτό. Ήταν σαφές λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα συμπορεύονταν. Συμφωνία λοιπόν σε πρώτη ανάγνωση. Αύριο ελπίζω όλοι μαζί, θα μπορέσουμε να βάλουμε τα θεμέλια για μια νέα συμφωνία θεμέλιο για περισσότερη διαφάνεια και περισσότερη ανταγωνιστικότητα των αγορών μας. Ας δούμε την οδηγία αυτή και μέσα στο πλαίσιο, στο κατάλληλο πλαίσιο. Ήδη τον Δεκέμβριο συντάξαμε την σχετική έκθεση για τα αγαθά εξοπλισμών. Πρόκειται τώρα για το δεύτερο βήμα που κάνουμε. Οι οδηγίες είναι βέβαια θεωρητικά ανεξάρτητες, στην πράξη όμως αλληλοεξαρτώνται. Και για το λόγο αυτό η ε, ψήφιση αύριο του πακέτου των εξοπλισμών είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν πρόκειται να προκαλέσει καμία επανάσταση στην αγορά. Είναι όμως σημαντικό βήμα πρόοδου και μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ευρωπαϊκή πολιτική αγορά εξοπλισμών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω του συναδέλφου μου, την κυρία Σολότε Σέντερσιολτ, ε, και τις άλλες οι ε, σκιώδεις εισηγητές που με συνόδευσαν με κριτικό πνεύμα αλλά πάντοτε ε, διαθέσιμες για συνεργασία. Για όλους τους συμμετέχοντες και εδώ, ενώ εδώ και τους εκπροσώπους των άλλων θεσμικών οργάνων όλοι συνεργάστηκαν γιατί είναι σημαντικό να γίνει μια συνεργασία το οφείλουμε στους πολίτες, στους Ευρωπαίους πολίτες και ελπίζω αύριο να ολοκληρωθεί αυτή η συνεργασία με την υπερψήφιση του πακέτου αυτού. Κατά τα άλλα θεωρώ ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει στις Βρυξέλλες και όχι στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ κύριε Λάμστροφ. Ο ε, Επίτροπος κ. Μακρύβη. Αξιότιμοι βουλευτές, σας ευχαριστώ. Συμπαθήστε με και για την φωνή μου, αλλά είμαι λίγο κρυωμένο. Έχουμε αυτό το σχέδιο οδηγίας που αφορά αυτές τις συμβάσεις προμήθειας παραγής υπηρεσιών. Είναι αυτό το λεγόμενο πακέτο για την άμυνα. Πρόκειται για τη γνώμη μου για ένα θετικό βήμα, ούτως ώστε να έχουμε μια αγορά κοινή και στον τομέα της άμυνας. Αυτό θα βοηθήσει για την πολιτική μας, την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Πολύ σημαντικό θα αναβαθμιστεί η αμυνά μας, θα θωρακιστούν οι δαπάνες μας. Έχουμε μια διαδικασία διαπραγμάτευση που προηγήθηκε, ε, έγινε στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Και ευχαριστώ επ' αυτού τον κύριο Λάμστρουφ που εντατικά και αποτελεσματικά δούλεψε ούτως ώστε σε πρώτη ανάγνωση να πετύχουμε μια συμφωνία. Οι δε και αυτοί συνεργαστήκανε επικοδομητικά μαζί μας αλλά βοήθησε πολύ η, Σλο... Σλοβενική συγγνώμη, και Γαλλική Προεδρία. Καθόλου στις διαπραγματεύσεις ή στο Συμβούλιο. Τέλος, πρέπει να πω ότι βοήθησε ιδιαίτερος και η Τσεχική Προεδρία. Νομίζουμε ότι είναι κομμένη και ραμμένη αυτή η οδηγία στι ανάγκε ε, τη ασφάλεια και τη άμυνα όσον αφορά αυτέ τι συμβάσει που πολλέ φορέ ε, είναι ε, για θέματα λεπτά, ευαίσθητα, πολύπλοκα. Βεβαίω και εδώ υπάρχουν και θέμα διαφανών πληροφοριών και υπάρχει και εξασφάλιση για κάθε προμήθεια. Αυτό ελπίζουμε να βοηθήσει τα περισσότερα κράτη-μέλη όσον αφορά τις συμβάσεις στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας. Μιλούμε για προμήθειες που αφορούν πολύ σημαντικά, λεπτά θέματα. Είναι θέματα πραγματικά στρατηγικά, για κάποιες απειλές υπερεθνικές. Και πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με υπέρβαση της γραμμής που χωρίζει τις ε, αστικές υποθέσεις, ας τις πούμε, από τις στρατιωτικές. Και μιλούμε για υλικό άμυνας και συναφές που εξομοιούνται με λίγο αμήνους. Με αυτή την οδηγία τα άρθρα, τα συγγνώμη, κάποια κρατημέλη να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια παρέκκληση που προβλέπεται δυνάμει το άρθρο 296 συνδίκης για Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι ελπίζουμε να υπάρχει διαφάνεια, να υπάρχουν υγιείς συνθήκες ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές. Θα ωφεληθεί και η βιομηχανία, η παραγωγή, οικονομίες κλίμακας θα έχουμε. Έτσι πιστεύουμε ότι οι δαπάνες θα συγκρατηθούν και οι τιμές θα δημορφωθούν με τέτοιο τρόπο που να ωφεληθούν όλοι. Και έτσι επίσης θα έχουμε περισσότερο value for money, θα πιάσουν τόπο τα χρήματά μας. Και η επιτυχία μας οφείλεται κατά πολύ στο έργο το οποίο επιτελέσατε και πάλι ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα η κυρία Σέντερσουλ για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ. Εδώ δεν μπορούμε να φτιάχνουμε μέσα στη νύχτα, μέσα σε μια νύχτα την ενιαία αγορά για τα θέματα των, ε, Όχι. της άμυνας και της ασφάλειας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει φυσικά και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας και των Ρωτών που είμαι μέλος. Είναι θέμα της των αρμοδιοτήτων μας βέβαια το θέμα αυτό. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε τι κατάλληλε συνθήκε, γιατί το μέσο αυτό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει κάνει και η γαλλική κυβέρνηση πολλά, αλλά πάνω από όλα ο κύριο Λάμστορφ, ο εισηγητή ήταν αυτός που συνέβαλε τα μάλα στην εξέλιξη του προγράμματος των ε, προτάσεων και Πιστεύω ότι θα πρέπει και η οδηγία ε, για τις ε, προμήθειες του 2004 να ληφθεί υπόψη στην υπόθεση αυτή. Και επίσης έχουμε και θέματα τόσο εθνικής ασφάλειας, όσο, εθνικών συμφερόντων θέλετε, όσο και ασφάλεια στη διακίνηση των προμηθειών, αλλά και των πληροφοριών Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, ισχύσει το άρθρο 296 όπου ε, αρμόζει, αλλά βεβαίως χωρίς καταχρήσεις. Και να έχει τη δυνατότητα και η βιομηχανία μας να αναπτύσσει νέες ε, σύγχρονες πρακτικές. Με χαρά βλέπουμε ότι το Συμβούλιο ανταποκρίθηκε σε κάποιες από τις ανησυχίε που είχαμε εκφράσει για τα όρια επί για το κατόφλι δηλαδή, αλλά και για θέματα διαφάνειας ένα από τα παραδείγματα μόνο των επιτυχιών που σημειώσαμε. Προσωπικώς δε βλέπαμε χαρά ότι τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα βρήκαν απαντήσεις χάρη ή μπορούν να βρουν απαντήσεις χάρη στην υφιστάμενη, στην ήδη ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο λοιπόν υποστηρίζει την ε, έκθεση με βρήτατη πλειοψηφία ελπίζουμε και θα σημάνει με την συμπεριφορά του αυτή ένα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου. Χαίρομαι και ευχαριστούμε πολύ όλους τους συναδέλφους για την επικοδομητική συνεργασία στο σημαντικό αυτό θέμα. Ο κύριος Βάιλερ, ξανόμενος των Σοσιαλιστών, για τέσσερα λεπτά. Κύριε Βάιλερ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Με το νέο χρόνο είχαμε μεγάλες, μεγάλους πηχαίους τίτλους για την, για τους εξοπλισμούς, για τον ανταγωνισμό στους εξοπλισμούς, για τη διαφθορά σε θέματα τέτοια, τόσο στη Γερμανία όσο και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν για εμάς τους ευρωδημοκράτες είναι σαφές ότι αυτοί οι εξοπλισμοί, ο αγώνας δρόμου για τους εξοπλισμούς αλλά και τα προβλήματα της διαφθοράς που συνδέονται με τα θέματα αυτά είναι καταδικαστέα από όλους εμάς τους Ευρωπαίους Ελληνοκράτες. Οι δύο οδηγίες λοιπόν μεταφορές και αναθέσεις θέλουμε να προχωρήσουν μόνο όταν είμαστε βέβαιοι ότι δεν κινδυνεύουμε από διασπάθηση χρημάτων δημοσίων, το χρημάτων δηλαδή του Ευρωπαίου Φορολογουμένου, όταν δεν γίνεται αγώνας δρόμους εξοπλισμένους, ποιος θα πάρει πες τώρα όπλα, και μόνο τότε μπορούμε να δώσουμε στους δημοκράτες την ε, ε, ψήφο υποστήριξής μας. Όταν μπορούμε να ε, υπηρετήσουμε την άμυνα και την ασφάλειά μας. Βεβαίως, θα πρέπει να προχωρήσουν αυτές τις λύσεις με περισσότερη συνεργασία όμως μεταξύ των κρατών μελών, χωρίς επικάλυψη των προσπαθειών, χωρίς προσπάθεια να ικανοποιηθούν μόνο τα συμφέροντα της, των βιομηχανιών όπλων. Για μας, τους ευρωβουλευτές, και, πάνω, και εδώ μιλώ από όλες τις ομάδες πιστεύω, κύρια σημασία ήταν η πρόταση της κυρίας Φουρτού με την οδηγία οι κυρώσεις σε περιπτώσεις διαφθοράς ή προβλημάτων να φτάνουν μέχρι και τον αποκλεισμό από ανάθεση συμβάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο και τελικά μπορέσαμε να το επιβάλλουμε, ελπίζω, ε, και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα αυτά θα είναι αποτελέσματα αποδεκτά και βιώσιμα για τα 27 κράτη-μέλη, έστω και είναι μόνο λίγα αυτά τα οποία έχουν δική τους ζωμηχανία όπλων. Είναι απαραίτητο και τα 27 κράτη-μέλη να συμπράξουν στην υπόθεση αυτή. Βλέπω ότι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής. Δεν είμαι μόνο βέβαιη για το κατά πόσον θα λειτουργήσουν τα πάντα όπως θα θέλαμε. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει, και το έχουμε συμπεριλάβει αυτό στις προτάσεις μας, να συμπράξει και να είναι σε θέση να παρακολουθεί την κατάσταση και μετά και να ελέγχει, όχι κατά τρόπο αυτοματοποιημένο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά να μπορούμε να επαληθεύουμε τα αποτελέσματα και τον τρόπο λειτουργίας αυτής της οδηγίας, αυτού πακέτου καλύτερα, και όταν στο μέλλον έχουμε μια ισχυρότερη αγορά, εσωτερική αγορά, θέλουμε να έχουμε και περισσότερες αρμοδιότητες, όπως άλλωστε έχει ήδη προβλεφθεί, και Ελπίζουμε ότι θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι εκείνο το όργανο με τους αιρετούς εκπροσώπους των πολιτών, το θεσμικό αυτό όργανο, το οποίο θα μπορεί να ασκήσει ουσιαστικό έλεγχο σε αυτέ τι συμβάσει. Όπω γίνεται άλλωστε από τα εθνικά κοινοβούλια, είναι αρμοδιότητα των εθνικών κοινοβουλίων και μια αρμοδιότητα που διεκδικεί το κοινοβούλιο στο, για το μέλλον. Εμεί οι Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτε με την ε, βιομηχανία όπλων με πολύ υψηλέ τιμέ και κόστο στα μεγάλα σχέδια που αναπτύσσουμε. Ε, έχουμε βέβαια αδυνατή εμπειρία του ελέγχου του κοινοβουλευτικού στι συμβάσει αυτέ και ίσω να υπάρχουν και οι λοιποί συνάδελφοι από τα άλλα κράτη-μέλη αντίστοιχη εμπειρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία. Τα αποτελέσματα ήταν καλά. Βλέπω πάντω ότι ορισμένα προβλήματα δεν μπόρεσαν να αντιμετωπιστούν όπως θα θέλαμε γιατί οι συμβιβασμοί σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή δεν είναι σωστή κοινοβουλευτική δουλειά και θα θέλαμε αυτού του τύπου οι διαδικασίες, ή οι λύσεις να χαρακτηριστούν, να είναι μόνο μια κατεξαίρεση ε, επιλογή και να μην δούμε να επαναλαμβάνεται συχνά γιατί δεν θέλουμε να καταργηθεί το πραγματικό κοινοβουλευτικό έργο και λειτουργήμα. Ευχαριστώ, Ο κύριος Μπουσόη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο κύριο Λάμπστορπ για την εξωτερική έκθεση. Ξέρω ότι ήταν πολύ αφοσιωμένο στη δουλειά του, ήταν εξαιρετική ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο για την κοινή αγορά πώληση ε, των ε, αμυντικών εξοπλισμών και χαιρετίζω ότι οι αρχές της συνθήκης, η μη διακριτική μεταχείριση και η διαφάνεια θα εφαρμοστεί και στην αγορά αυτή των όπλων και αυτό θα, είναι ακριβώς, θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των αμυντικών δαπανών. Ο συνάδελφος, ο κύριος Λάμστορφ, ε, παρουσιάζει κάποιες ε, αρχές που θα επιτρέψουν να λειτουργήσουν σωστά ή, να λειτουργεί σωστά η κοινή αγορά των όπλων. Θα ήθελα σωστα η κοινη αγορα δύο βελτιώσεις αν θέλετε και για τους ε, παραγωγούς αλλά και για τις αναθέτουσες αρχές όπου θα βελτιώσει την ασφάλεια των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια προμηθειών θα πρέπει να έχουμε λεπτομέρειες για τους παραγωγούς και για τους ενδιάμεσους και θα πρέπει οι αναθέτουσες αρχές να εξασφαλίσουν μια σωστή πληροφόρηση και από την άλλη πλευρά οι δημοπράτες θα πρέπει να εξασφαλίζονται από, την, από σαφείς διαδικασίες έτσι ώστε να μην, υπάρχουν, να υπάρχει διακριτική μεταχείριση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τα συμφέροντά τους, κυρίως χορηγώντας, μη χορηγώντας εξαιρέσεις όσον αφορά την... Ε, μάλλον εξαιρέσεις όσον αφορά την... Ε, ε, το ότι πρέπει να δίνουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες σε περίπτωση που απειλείται η δημόσια ασφάλεια στο μέλλον, εάν εξετάσουμε κάπου πιο, πιο ευαίσθητα θέματα πέραν της αγοράς ε, όπλων, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την, ε, το στρατηγικό συμφέρον κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστώ ο κύριος Γιανόφσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Λάμστορφ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και κυρίως όσον, γιατί όσον αφορά τα, τις δημόσιες δαπάνες ε, είναι ένας τομέας που όλους μας ενδιαφέρει και εδώ είναι ακόμα πιο ευαίσθητο το θέμα, μια και μιλάμε για τις αμυντικέ δαπάνες, μιλάμε για τεράστια ποσά, θα πρέπει να επιλέξουμε συγκεκριμένους προμηθευτές που θα μας προσφέρουν όχι μόνο την πιο φτηνή λύση αλλά και την ε, βέλτιστη θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και την ισότητα ε, των εργαζομένων, τον, ε, την, ότι πρόκειται για τη σωστή εργασία και υπάρχουν και θέματα απορρίτου τα οποία πρέπει να σεβαστούμε σε ορισμένες ε, περιπτώσεις. Επίσης, όσον αφορά τα αντισταθμιστικά, ε, ωφέλη. Ε, η θέση η οποία παρουσιάζεται στο σχέδιο είναι πάρα πολύ σωστή. Θα πρέπει ε, να βάλουμε ένα πλαίσιο, αν θέλετε, στις αμυντικές δαπάνες. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ευχαριστώ πολύ, πολύ. Καλή ήταν η συνεργασία και ο εισηγητή έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και παρά τις επικρίσεις προς τη διαδικασία για την πρώτη ανάγνωση ήταν προϋπόθεση όλη αυτή η καλή συνεργασία ώστε να ε, ληφθεί υπόψη πράγματι η θέση του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο ουσιαστικά. Σήμερα λοιπόν ε, καλούμεθα να συζητήσουμε ένα συμβαστικό προϊόν διαπραγματεύσεων θα έλεγα σε μια σε ένα τομέα όμω που ήταν αποκλεισμένο από την εσωτερική αγορά μέχρι τώρα και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για μένα το να βλέπω την αντιπαράθεση που είναι οικία στον τομέα τη εσωτερική αγορά ε, και τη προστασία των καταναλωτών να εφαρμόζεται σε θέματα εξοπλισμών κτλ. και άμυνα. Πολύ καλό λοιπόν αυτό, πολύ, πολύ καλή εξέλιξη και γιατί. Γιατί όταν έχουμε να κάνουμε αμυντικά συστήματα και προϊόντα και πρέπει αυτά να κριθούν με κριτήριο και τις τιμές εξασφαλίζουμε πιο αποτελεσματική χρήση του δημόσιου κορβανά πράγμα το οποίο βέβαια ισχύει και για τον περιορισμό των φαινομένων διαφθοράς που οφείλουμε να επιτύχουμε για χάρη του πολίτη της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα δικασίες που επιτρέπουν τις συνθήκες εκείνες για πιο καλό ανταγωνισμό, που θα δώσουν και μια ευκαιρία ανταγωνιστική στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μειώσουμε τα διάφορα παραθυράκια ε, που θα επέτρεπαν σε κάποιον να αποφύγει τη δημόσια προκήρυξη και σε αυτό θα πρέπει βέβαια να επικοινωνούμε και να συνεργαζόμαστε και με την Επιτροπή και Μπορεί μέχρι τώρα να απαγορεύονταν ε, νομοθετικός πόσει, το γράμμα τουλάχιστον του γρόμου του νόμου, ε, τώρα βλέπουμε ότι μπορούμε να απορρίψουμε τέτοιες πρακτικές και εν τέλει μπορούμε να προβλέψουμε και ένδικα μέσα στις διαδικασίες αυτές των διαγωνισμών των δημοσίων προμηθειών. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι προχωρούμε προς περισσότερη διαφάνεια. Ίσως να μην έχουμε πετύχει το στόχο μας ακόμη, την απόλυτη διαφάνεια, αλλά πάντως εδώ έχουμε να κάνουμε ένα σημαντικό ορόσημο. Ευχαριστώ ο κύριος Φλούγκερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μέρος ε, του πακέτου για την άμυνα, με τον δική αυτή, υποτίθεται ότι θα βοηθήσουμε για μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία αμυντικών, ε, την αμυντική βιομηχανία στην Ευρώπη. Δηλαδή για, για εξοπλισμούς, δηλαδή για όπλα, που είναι βέβαια η πηγή κάθε καταστροφής με τον πόλεμο. Άρα τι θέλουμε, να έχουμε τους καλύτερους εξοπλισμούς στην Ευρώπη. Ο κύριος Φόποντα το έφερε αυτό το θέμα λίγο πολύ στην ομιλία του. Είπε δηλαδή ότι η βιομηχανία των εξοπλισμών θα βρίσκεται σε καλή θέση εναντί των ανταγωνιστών της κυρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 2005 ήταν η πρώτη φορά όπου ε, χαρακτηρίστηκαν ε, ως πρώτοι σε εξαγωγές ε, οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι όπλων. Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία ήταν οι πρώτοι των πρώτων με κύριους αποδέκτες στη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια πιο ανταγωνιστική ή πιο αποτελεσματική οπλική βιομηχανία. Ο μας θα έπρεπε να είναι ο αφοπλισμός και όχι η ανταγωνιστικότερη μηχανία των όπλων. Ξέρουμε πάρα πολύ τι νόημα και τι σκοπό έχει αυτή η οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. ΣΠΑΠ για τρία λεπτά. Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τι ευχαριστίε μου προ την Επιτροπή ε, τη Ιστορική Αγορά και τη Προσφυγή των Καταναλωτών, αλλά και προ τον εισηγητή ιδιαίτερο τον ε, κύριο Λάμστορφ αλλά και τον πρόεδρό της, ε, τον κύριο Φολφόγκαο που μας έχει τόσο πολύ βοηθήσει σε αυτήν την υπόθεση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το ζήτημα όχι το πόσα όπλα θα παράγονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πολλούνται εκτός αυτής, αλλά το υπό ποιες συνθήκες θα διατίθενται ή, ε, τα συστήματα αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα 27 κράτη-μέλη, υπό συνθήκες διαφάνειας και βέβαια πολύ χαμηλότερων τιμών. Πιο πρακτικά δηλαδή ζητήματα και γι' αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να χαιρετήσω εκ μέρου και των πολιτών αυτή την προσπάθεια για μια μεγάλη αγορά, μια αγορά των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο που θα μπορέσει να δει Μεγάλε μεγάλες οικονομίες και πολύ πιο αποτελεσματική λειτουργία. Πρόκειται για μια συνεργασία και βέβαια λυπούμε που δεν είναι καλύτερη εκπροσώπηση του Συμβουλίου σήμερα στη συζήτηση. Η απόφαση λοιπόν αυτή ιδιαίτερα πρέπει να χαιρετηθεί και γιατί. Γιατί είχαμε πολύ μεγάλε δυσκολίε στι ε, συνομιλίε και την ε, προσπάθεια για την διαπραγμάτευση μεταξύ κρατών μελών στο παρελθόν. Τώρα όμω με τον τριμερή διάλογο και με την ε, ισότιμη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων βλέπω ότι μπορούμε να αναπτύξουμε το όραμα για μια ουσιαστική πολιτική άμυνας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Ε, βλέπω με λύπημα ότι είναι πολύ λίγοι οι συνάδελφοι σήμερα εδώ στην Ολομέλεια. Σήμερα το πρωί που είχαμε την επέτειο των 10 ετών από την εισαγωγή του ευρώ ήμασταν επίσης πολύ λίγοι, δυστυχώς, αλλά ελπίζω ότι θα μπορέσουμε στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας να προχωρήσουμε πολύ καλύτερα γιατί στο μέλλον ξέρουμε πολύ καλά ότι οτιδήποτε μπορούμε να διεκδικήσουμε ή να ε, έχουμε σαν προσπάθεια σε ένα κράτος μέλος μπορεί να ισχύει και στα λοιπά. Και γι' αυτό μπορούμε να έχουμε πολύ καλέ ελπίδε για το μέλλον. Ευχαριστώ ιδιαίτερω λοιπόν για την έκθεση αυτή και ιδιαίτερα ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία τη στην υπόθεση αυτή και ε, χάρη στην οποία μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε όποια προβλήματα είχαμε σε σχέση με ορισμένα κράτη-μέλη και έτσι μπορέσαμε να βοηθήσουμε και το, και το Κοινοβόλιο στην ε, προσπάθεια εισαγωγή πιο αυστηρών διατάξεων ω προ την ε, νομοθεσία που ισχύει, που για τους ε, διαγωνισμούς, για τις αναθέσεις. Το δεύτερο ζήτημα που έχει να κάνει με την ένταξη στον τομέα της εσωτερικής αγορά των αμυντικών συστημάτων της αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα θέμα το οποίο ιδιαίτερα θα πρέπει να χαιρετήσουμε, ένα θέμα το οποίο οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό και στις προσπάθειες των συναδέλφων της Επιτροπής Ιστορική Αγορά και ε, Θεμάτων του Καταναλωτή. Όταν έχουμε λοιπόν ε, τη δυνατότητα να αποστέλουμε στρατεύματα σε διάφορες περιοχές του κόσμου για να ε, βοηθήσουμε στην ειρήνευση, σημειώνουμε ότι είναι μεγάλη καθυστέρηση προ τη δημιουργία μια Ευρωπαϊκή Ένωση τη Άμυνα. Και σε αυτό έχουμε καθυστερήσει και θα πρέπει να προχωρήσουμε το δυνατόν πιο γρήγορα. Ευχαριστώ. Κύριο Φεραίρα. Πρώτα-πρώτα, Πρόεδρε, στον ε, εισηγητή του κ. Λάμπτορ αλλά και στου ε, εισηγητέ, του σκιώδη, θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια και φυσικά ξεχωρίζει εδώ ο ρόλος της Μπάρμπαρα Βάιλερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι πολύ σωστό να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά την, τον συντονισμό, τον στρατηγικό συντονισμό των παράγοντων μας. Θα πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα μπρος, τόσο ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει με τις βιομηχανίες άμυνας. Θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια σε αυτές τις, ε, στους διαγωνισμούς, αλλά και στις συμβάσεις που τελικά συνάπτονται. Ε, επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε ε, να δούμε πώς θα έχουμε ανταγωνιστικότητα στα ε, ευρωπαϊκά προϊόντα στις παγκόσμιες αγορές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Πρόεδρε, με αυτή την οδηγία να μπορέσουμε να κάνουμε κατά προς όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στο οποίο κινούνται οι δημόσιες συμβάσεις για την ασφάλεια και την άμυνα. Ε, πρέπει φυσικά να σεβαστούμε τα συμφέροντα των κρατών μελών και κυρίως ε, τα συμφέροντα ε, που αφορούν την ασφάλεια αλλά και ε, την βιομηχανία όπλων και γενικά εξοπλισμού άμυνα και ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε ότι δημιουργούνται συνθήκες ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ε, καλύτερη προσβασιμότητα εκ μέρου των ΜΜΕ στην αγορά, ε, γιατί έχουν βελτιωθεί οι κανόνε σχετικά με την υπεργολαβία και με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατόν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να έχουμε μια αυθεντική αγορά στην Ευρώπη για του τομεί αυτού άμυνα και ασφάλεια και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε και όσον αφορά την ε, έρευνα για όλες ε, τις ε, βιομηχανίες στην Ευρώπη να τις βοηθήσουμε. Για όλες αυτές οι οποίες συμμετέχουν στα θέματα της άμυνας. Τέλος, συνάδελφοι, θα πρέπει να αναφέρουμε το πώ θα αναπτυχθούν οι βιομηχανίε που έχουν σχέση με την άμυνα και εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση εν κατακλείδη, θα πρέπει να σα πω ότι να μην ξεχνούμε την ρίση ότι όποιο θέλει ειρήνη θα πρέπει να προετοιμάζεται για τον πόλεμο. Είμαστε μια με μια ειρηνική δύναμη. Όμω είναι σημαντική η προετοιμασία τη ε, άμυνάς μας για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη. Ο έχετε ένα λεπτό κύριε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω να σας πω τα εξή Μιλούμε για 500 εκατομμύρια δολάρια τα οποία δαπανώνται στην έννοια του Ατλαντικού για ασφαλεία και άμυνα. Εμείς βρισκόμαστε στα 200 Οπότε το ερώτημα αναδύεται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα 200 δις και να φτάσουμε πολεμική ικανότητα και αμυντική όπως η είπα έκανα Υπουργό Άμυνα. και τότε συνάντησα εκπροσώπους της σχετικής βιομηχανίας. Και του είπα, είμαι υπουργό άμυνα, τους είπα τότε, αλλά δεν είμαι υπουργό που αμήνεται υπέρ τη βιομηχανία σα. Ε, Βεβαίω ο κύριο ε, Λάμστορφ ε, έκανε αυτή την έκθεση και η οδηγία πρέπει να δεχθούμε ότι μα βοήθησε ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πιο ορθολογική δαπάνη των πόρων μα και έτσι θα βελτιωθεί η αμυντική ικανότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, να πρέπει να έχουμε αμυντική ικανότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, ο κύριο Μπέιρ. Κυρία Μπέιρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφοι, θα ήθελα να υπογραμμίσω τέλο ότι έχουμε να κάνουμε με μία λύση, σε μία δέσμη μέτρων. Αυτό είναι το θέμα που συζητούμε σήμερα με όλη αυτή τη συζήτηση και για την οδηγία για τις ε, δημόσιες σε όπλα για τις συμβάσεις. Στόχος μας είναι με την αναρμόνιση της ε, ε, βιομηχανίας των εξοπλισμών στην Ευρώπη να έχουμε ισχυρότερο έλεγχο μαζί βέβαια με την ένταξη στην εσωτερική αγορά αυτών των ε, αγορών, αυτών των συμβάσεων, να έχουμε καλύτερο έλεγχο. Γι' αυτό με εκπλήσουν οι αντιδράσεις που ακούω από ορισμένους στο Συμβούλιο τελευταία χρόνια, στις τελευταίες συνεδριάσεις, στο τελευταίο χρόνο καλύτερα υπό τη Γαλλική Προεδρία, υιοθέτησε τον κώδικα καλή συμπεριφοράς, όπως άλλωστε στο το Κοινοβούλιο παγίως. Αυτό θα ήθελα ιδιαίτερω να υπογραμμίσω ότι η εναρμόνιση αυτή την οποία θεωρούμε θετική εξέλιξη υπάγεται στον έλεγχο των κρατών μελών και μάλιστα όχι μόνο η εναρμόνιση αλλά και η επεξεργασία των μηχανισμών κυρώσεων για την περίπτωση των παραβάσεων στις διατάξεις της ε, οδηγίας. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Στουμπών για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο συνάδελφος κ. Βάμπ πριν από λίγο. Πρέπει να σας πω ότι η υιοθέτηση σήμερα αυτής της οδηγία είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και την οφείλουμε στις προσπάθειες του εισηγητή μας, του κ. Λάμπστορφ, της, ε, του σκιώδη εισηγητή Σιόντρου Σόρφο και στην ε, Γαλλική Προεδρία που στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να καταλήξουμε σε μια συμβαστική λύση. Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι να ολοκληρώνουμε έναν κύκλο ο οποίος ήταν πάρα πολύ γρήγορος, κράτησε μερικούς μήνες που, που περιλαμβάνει και την ε, έκθεση για τα ε, για τις αμυντικές ε, αγορές ε, το Δεκέμβριο, τον κώδικα συμπεριφοράς και αυτήν εδώ την οδηγία που έχει σαν στόχο να συμφιλιώσει το άρθρο 296 της συνθήκης με τους κοινού κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις. Όλο αυτό το σύνολο ουσιαστικά, επιτρέψτε μου να πω, ότι μας δεσμεύει να κοινοτικοποιήσουμε την αγορά της άμυνας. Αυτό ενδεχόμενα να εμφανίζεται ερετικό σε σχέση με τις απαιτήσεις ε, για κυριαρχία και με βάση τα ε, κύρια χαρακτηριστικά της αμυντικής πολιτικής. Αυτό εκφράζει μια ε, προσπάθεια ολοκλήρωσης σε αντίθεση με τις εθνικές κυριαρχίες και κατά διάρκεια της γαλλικές της Γαλλικής Προεδρίας αλλά και η Πορτογαλική και η Σλοβενική Προεδρία κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες σε έναν τομέα όπου οι εθνικές κυριαρχίες θεωρούσαν ή ε, ε, μας ανάγκαζαν να Πιστεύουμε ότι δεν θα καταλήγαμε σε οποιαδήποτε συμφωνία. Πιστεύω, Πρόεδρε, ότι με το κείμενο αυτό εδώ ε, ολοκληρώνεται η συζήτηση για την φύση ε, της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σημαντική δύναμη ε, και αυτή θα εμφανιστεί και στην αμυντική πολιτική και στην εξωτερική πολιτική. Ο κύριος Βανόρντεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ε, οι Βρετανικοί συντηρητικοί ε, ε, υπεραμεινόμεθα της ελεύθερης ανοιχτής αγοράς. Όμως όπως είπαν πάρα πολλοί ομιλητής το κείμενο αυτό δεν οδηγεί σε κάποιο οικονομικό συμφέρον απλώς ολοκληρώνει περισσότερο την ενιαία αγορά. Δεν βελτιώνει ούτε καν τις αμυντικές ικανότητες και σε σχέση Υπάρχουν, ε, παρουσιάζει όμως ε, πλεονεκτήματα και για την δίσδυση βρετανικών προϊόντων σε άλλες αγορές αλλά και το ανάποδο και η βρετανική αγορά είναι πιο ανοιχτή στην Ευρώπη. Το πρόβλημά μας είναι ότι σύμφωνα με τις προκινόμενες ε, ρυθμίσεις κάποιες δαπάνες δεν θα επιτρέψουν ε, να ε, ανακτήσουμε τις, ε, τα χρήματα αυτά στην φάση ανάπτυξης οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα μπορέσουν να διαφυλάξουν ούτε την πνευματική ιδιοκτησία, ούτε την ασφάλεια των θέσεων απασχόλησης. Και υπάρχουν και άλλες ανησυχίες, Πρόεδρε, αλλά πρέπει να σας πω ότι η έκθεση αυτή δεν είναι απολύτως απαραίτητη από πλευράς αμυντικής, βιομηχανικής ή οικονομικής σκοπιάς. Ο κύριος Πάσκο για ένα λεπτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της, ε, της, της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Όντως θα πρέπει οι, δαπάνες, οι, οι συμβάσεις αυτές να ε, λαμβάνουν υπόψη και το θέμα του, του απορρίτου ε, και υπάρχουν δύσκολοι κανονισμοί και λεπτομέρειες ε, οι οποίες είναι δύσκολες, συμφιλιώνονται πάρα πολύ δύσκολες ε, να γίνουν σεβαστές διότι θα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας και την διακριτικότητα και το απόρριτο και τη διαφάνεια επομένως θα πρέπει να γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την ισορροπία ανάμεσα σε όλες αυτές τις αξίες. Θα πρέπει ε, οι αρχές της κοινότητας να παίζουν το ρόλο διαιτητή σε αυτή την ε, αγορά που δημιουργείται ε, και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Μια, αυτές αυτοί οι κανόνες όμως για κάποιες χώρες όπως ε, η Ρουμανία ε, είναι απαραίτητες για την ε, διάσωση της εθνικής μας βιομηχανίας. Ο κύριος Μαρινέσκου. Πρόεδρε, η οικονομική κρίση έθεσε σε κίνδυνο, όπως και η ενεργειακή κρίση, την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαπιστώσαμε όμως για άλλη μια φορά ότι μόνο χάρη στην Ένωση και την ενότητα μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή και την ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες κρίσεις ε, που αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο προβλήματα της ασφάλειας ε, και η νέα αυτή οδηγία είναι ένα βήμα προόδου για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί προβλέπονται διαδικασίες ε, κατάλληλες, διατυπώσεις σωστές έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι αναθέσεις, οι δημόσιες ε, συμβάσεις κατά τρόπο ουδέτερο αντικειμενικό και για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τους μεγάλους ανταγωνισμούς μας και ιδιαίτερα των ΗΠΑ. Χρειαζόμαστε τον έλεγχο των εξαγωγών των προϊόντων στον τομέα της άμυνας προς χώρες τρίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, με την κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας, θα, σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, θα μπορέσουμε να έχουμε μια διαρθρωμένη και διαρκή ε, συνεργασία στον τομέα αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Λογκάνσκι. Πρόεδρε, είδαμε τον κατακαιρματισμό των ε, αμυντικών μηχανιών στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 60 και μετά με αποτέλεσμα να ε, αυξάνονται οι δαπάνες, να μειώνεται η αποτελεσματικότητα και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Τώρα όμως για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε το κατάλληλο, το απαραίτητο στρατικό δυναμικό στα κρατημέλη χρειάζομαστε τεχνολογία, τεχνολογική βάση, έρευνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι μεγάλε προκλήσει στο μέλλον, στον τομέα τη ασφάλεια. Επίση, θα πρέπει να έχουμε ένα νομικό πλαίσιο πιο ομοιόμορφο που θα επιτρέπει και στα κράτη-μέλη την εφαρμογή των ευρωπαϊκών διατάξεων χωρίς να υπονομεύονται το, το, το, το, δυναμικό για άμυνα που μπορεί να έχει το κάθε κράτος μέλος. Και θέλουμε βέβαια και ουδέτερη αντικειμενική διαδικασία, ασφαλή, χωρίς ε, διακρίσεις. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον συντάκτη της έκθεσης, τον κύριο Λάμπστορφ, αλλά και ταυτόχρονα και τους σκιώδεις που έκαναν σπουδαία δουλειά. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς είναι ο κατακαιρματισμός που επικρατεί σε εθνικό επίπεδο η εξαγωγή προϊόντων συνδεωμένων με τον εν λόγω τομέα της άμυνας και της ασφάλειας υπόκειται σε εθνικά συστήματα αδειοδότησης που διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη διαδικασία το πεδίο εφαρμογής και τις προθεσμίες. η νέα αυτή νομοθεσία προωθεί τη διαφάνεια και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας ανοιχτής ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού που αποτελεί και βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. είναι σημαντικό επίσης ότι προβλέπονται ε, σημαντικές διατάξεις διατάξεις για την ασφάλεια του εφοδιασμού και των πληροφοριών. αποσαφηνίζεται και η επίκληση του άρθρου δύο hundred and ninety των ευρωπαϊκών κοινοτήτων αλλά περιορίζεται πλέον σε πραγματικέ παρεκκλήσει όπω προβλέπεται από τη συνθήκη και όπω ζήτησε το ευρωπαϊκό δικαστήριο. Τέλο κλείνω σημειώνοντα ότι είναι σημαντικό ότι μέσω ευέλικτων ρυθμίσεων ενισχύεται ο ρόλο μικρομεσαίων επιχειρήσεων που για κάποια κράτη μέλη είναι κλάδο που απασχολεί χιλιάδε εργαζόμενου. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να συγχωρώ τον κύριο Λάμστροφ για το εξαιρετικό έργο το οποίο επέτέλεσε αλλά και τους κύριου και την κυρία Σέντοσελ ιδιαίτερος. Κάτι να σταθώ πάνω σε αυτό που είπε ο κύριο Τουμπών για το πόσο βοήθησε η Γαλλική Προεδρία ούτως ώστε να επιτύχουμε συμφωνία για την οδηγία. Όταν επανέλθουμε σε λίγα χρόνια φαντάζομαι τότε θα ε, συνειδητοποιήσουμε ότι δεν θα πρέπει να φοβόμαστε να μιλούμε για την ε, κοινή αγορά άμυνας γιατί αυτό είναι ένα κοινό μας συμφέρον. Είναι συμφέρον να υπάρχει άμυνα κοινή και να υπάρχει ανταγωνισμός στη σχετική αγορά. Είναι πολύ σημαντικό για πολλά κρατημέλη ε, αυτό το οποίο αναφέρεται αυτές οι ρυθμίσεις που υπάρχουν για την υπεργολαβία, συμβούλια και κομισιόν τελικά βοήθησαν να περάσει η θέση μας. Να υπάρχει δηλαδή για τις υπεργολαβίες περισσότερη διαφάνεια και μην υπάρχουν τέτοιες διακρίσεις επί τη βάση της προέλευσης του υπεργολάβου. Επίσης, τέλος, οι εθνικές αρχές να δικαιούνται να πάνε στο 30% όσον αφορά το, τη σύμβαση που συνάπτεται με τον υπεργολάβο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μακρύβη Επίτροπος έχει τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε, για το συμβασμό. Επίσης, θα πρέπει να δεχτούμε ότι έχουν πολλούς λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι. Μας βοήθησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα 17 Νοεμβρίου το οποίο ήταν το θεμελιό για αυτή την οδηγία. Επίσης, η τελική εκδοχή του κειμένου διαμορφώθηκε κατά πολύ από τις τροπολογίες της ε, Επιτροπής ΙΜΚΟ. Δεχόμαστε όλες τις τροπολογίες. Συμφωνούμε με όλα όσα θέλετε να πω σχέση με την τροπολογία. Νομίζουμε ότι έτσι θα κάνουμε τη διαφορά και ούτως να έχουμε μια αυθεντική αγορά στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη. Η αλήθεια είναι ότι πριν από πέντε χρόνια ήταν κάτι σαν επιστημονική φαντασία το να θεωρεί κανείς ότι θα υπάρξει μια τέτοια αγορά. Να που το όνειρο έγινε πραγματικότητα και άρα δεν μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μα για την ευκαιρία η οποία υπήρξε προ τούτο. Και τώρα, το λόγο έχει ο κύριο εισηγητή μα, ο κύριο Λάμστορφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Φανόρντε, θα σα θυμίσω ότι είστε ο μόνο ο οποίος υποστήριξε τι θέσεις τη άκρα αριστερά. Κύριε Φλίγκερ, εσεί είστε ο μόνο ο οποίο υποστηρίζει την άκρα δεξιά στις θέσεις σα ω προς την ιστορική αγορά. Για τόσο είπε η κυρία Βάιλερ θα ήθελα να πω ότι έχει δίκιο όταν λέει ότι πρόκειται για προϊόντα τα οποία χωρί ανταγωνισμό είναι πολύ ακριβά. Είναι πολύ ακριβά επειδή δεν έχουν ανταγωνισμό. Είναι για, ο λόγος αυτός για τον οποίο θέλουμε να δημιουργήσουμε μια ιστορική αγορά για τα προϊόντα αυτά, ώστε να είναι όχι φθηνιάρικα, αλλά πιο φθηνά πάντως, έτσι ώστε να δώσουμε μια μεγάλη ευκαιρία και για τη βιομηχανία μας ε, να ξανοιχθεί και προς νέες αγορές, να εισέλθει σε νέες αγορές, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και εμείς την ευκαιρία να εξασφαλίσουμε περισσότερη διαφάνεια για τον πολίτη μας, περισσότερες επιτυχίες δηλαδή για τον πολίτη, με μια πιο καλά διαρθρωμένη εσωτερική αγορά. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο νομίζω. Και κλείνοντα, θα ήθελα να σημειώσω προ του συναδελφού Χαραντόφ και Τουμπό ότι του ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία του σε αυτό το εγχείρημα εγχείρημα της δεύτερη, του δεύτερου πυλώνα, ενίσχυση δηλαδή, της πολιτικής ασφάλειας και άμυνα, αλλά ταυτόχρονα μέσω τη πρώτου, πρώτου πυλώνα, δηλαδή τη εσωτερική αγορά. Και ιδιαίτερα εξαιρετική ήταν η συνεργασία με τη Γαλλική Προεδρία, η οποία διαμεσολάβησε σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και χάρη σε αυτήν επιτύχαμε πάρα πολλά. Ήταν μεγάλη ευκαιρία αυτή για την Ευρώπη, την πολιτική της Ευρώπης, για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ευρώπης, για την Ευρώπη της ειρήνης και, της, ε, και των αξιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. <clears throat> επικαλούμε το 145 του κανονισμού, μια και αναφέρθηκε το όνομά μου με μια προσωπική αναφορά και θα ήθελα να μου δώσω την ευκαιρία να, μιλήσω. Οι χαρακτηρισμοί ως προς το ποιος είναι ο εξτρεμιστής εδώ νομίζω ότι μπορούν να ανταποδοθούν κυρίως αν κοιτάξουμε ποιος είναι ο εξτρεμιστής της εσωτερικής αγοράς. Εγώ είπα ότι μια ε, α, ένταση ως προς τους εξοπλισμούς, ως προς την εξο... αγορά των εξοπλισμών και τη βιομηχανία των εξοπλισμών θα οδηγήσει σε ένταση και των πωλήσεων όπλων και έξω από την Ευρώπη. Ε, η κλήγη η συζήτηση, η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη προχωρούμε στην ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή. Πρώτη ερώτηση κύριου Μπέργκα. 10 χρόνια ευρώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η εμπειρία που έχουμε από όλο το γενικότερο συντονισμό